ψηφίσουμε στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο θέμα είναι η έκθεση της κυρίας Ροδικράτσας Ευρωπούλου σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Προχωράμε καλά σήμερα και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι ενδεχομένω να υπερφορτώσαμε και τη συνάδελφο κυρία Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στην ε, Επίτροπο αν συμφωνεί. Πρόεδρε, με γνώστης πολλών θεμάτων φαίνεται απόψε. Κύριοι βουλευτές, κυρίες βουλευτές, από τον Απρίλιο του 2011 κάναμε σημαντικά βήματα προ τα εμπρό για να αναβιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δι μικρομεσαίων. Συζητούμε τώρα μέτρα στο πλαίσιο της πράξης για την εσωτερική αγορά. Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Είμαστε όμω πλέον δεσμευμένοι στην προσπάθειά μας να αναβιώσουμε, να επανεκκινήσουμε την εσωτερική αγορά. Δεν πρόκειται όμω μόνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εδώ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέε ευκαιρίε για επενδύσει και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη καθ' όλη την Ευρώπη. Οι ανάγκε είναι τεράστιε. Γνωρίζουμε τι ανάγκε των μικρομεσαίων όσον αφορά την χρηματοδότηση τη ρευστότητά του. Έχουμε δρομολογήσει διάφορα προγράμματα για εταιρείε που δεν είναι στο χρηματιστήριο και που εξαρτώνται αποκλειστικά από τι τράπεζε για χρηματοδότηση. Η υποδομή είναι ζωτική σημασία για την επανεκκίνηση τη οικονομία. Κάθε χρόνο μεταξύ 100 και 150 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύονται σε έργα υποδομή στην Ευρώπη. Σε άλλε τομεί όμω δεν υπάρχουν κεφάλαια για επενδύσει. Ο τομέας των κατασκευών είναι τομέας των οποίο οφείλουμε μεγάλο μερίδιο της απασχόλησης. Και εκεί οι επενδύσει κάθε χρόνο είναι γύρω στα 100 δισεκατομμύρια. Όμω η μακροχρόνια, η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση τη ανάπτυξη είναι κατακρεματισμένη και πολλέ φορέ οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει δεν βρίσκουν τα κεφάλαια που χρειάζονται. Έχουμε πολύ ψηλέ αποταμιεύσει στην Ευρώπη, όμω τα χρήματα δεν βγαίνουν προ την πραγματική οικονομία. Γι' αυτό και υποβάλλουμε την πρόταση για τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Το πλαίσιο που προτείνουμε αποσκοπεί στην δημιουργία μιας υποδομή, ενό μηχανισμού όπου τα κεφάλαια θα κυκλοφορούν ελεύθερα ανά την Ευρώπη χωρίς ιδιαίτερε απαιτήσει για τις επιχειρήσεις που τα χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή λιγότερα από 10 κράτη-μέλη έχουν νομοθεσία η οποία επιτρέπει σε τέτοια μακροπρόθεσμα κεφάλαια να λειτουργούν. Τα ΕΜΕΚ υπάρχουν αλλά υπάρχουν 50 διαφορετικοί τύποι τέτοιων ΕΜΕΚ και είναι δύσκολο οι επενδυτέ να επιλέξουν. Τα νέα ΕΜΕΚ, τα νέα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια και οι σχετικοί κανόνε θα διευκολύνουν τι επενδύσει σε μακροπρόθεσμα έργα τα οποία χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Εκ μέρου του Μισελ Μπαρνιέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευγνώμων στην κυρία Κράτσα και στους κοιόδης για την πρόταση αυτή. Επιλήθηκαν πολύ γρήγορα πολλά τεχνικά ζητήματα και έχουμε πλέον ένα πολύ καλό κείμενο μπροστά μας, το οποίο ανικατοπτρίζει και το πνεύμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να προωθήσουμε δηλαδή μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Και είναι και το πνεύμα της συνένεσης και του συμβασμού. Έχουμε στόχο, επαναλαμβάνω, την επανεκκίνηση τη οικονομία στην Ευρώπη. Το Κοινοβούλιο κατάληξε στο ίδιο συμπέρασμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται να κινητοποιήσουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των αποταμιεύσεων. Να ανοίξουμε τα κεφάλαια σε όλες τις νετές επενδύσεις. Να προσελκύσουμε όλους τους επενδυτές την λιανική αγορά και αυτό θα εξασφαλίσει και επιτυχία στην πρόταση αυτή. Επίσης, η ΟΣΕΚΑ. Η σημαντική επιτυχία των ΟΣΕΚΑ, των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητέ αξίες, αποτέλεσε ένα εξαιρετικό όχημα για επενδύσεις. Οι τροπολογίε τη Επιτροπή ΕΚΟΝ διευρύνουν το πεδίο των επενδύσεων έτσι ώστε να πηγαίνουν στο σωστό σκοπό. Διάβασα επίση την, την αναλυσή σα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε ακόμη αντιμετωπίζουν δυσκολίε χρηματοδότηση. Δεν έχουμε αντίρρηση να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή τη πρόταση και να διευκολύνουμε και αυτέ. Όμω δεν μην ξεχνούμε ότι ο βασικό στόχο μα είναι οι επιχειρήσει και οι επενδύσει που χρειάζονται μακροπρόθεσμε επενδύσει, όχι όμω τι πολυεθνικέ επιχειρήσει. Απαιτούμε επίση ένα ελάχιστο ποσοστό επιχειρήσεων και επενδύσεων να είναι στην Ευρώπη. Διότι, παραλαμβάνω, οι επενδύσει που χρειαζόμαστε είναι επενδύσει στην ευρωπαϊκή οικονομία. Φυσικά έχουμε μια υποχρέωση. Όλοι μα οι νόμοι να συμβάλλουν με την συνθήκη. Γι' αυτό και οι νομικέ μα υπηρεσίε εξετάζουν κατά πόσον ε, κάτι τέτοιοι κανόνε είναι δυνατοί. Το πιο σημαντικό όμω σήμερα απόψε είναι το Κοινοβούλιο να προχωρήσει και να εγκρίνει το κείμενο, διότι ο τελικό στόχο είναι να βοηθήσουμε τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή οικονομίας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα είναι ει βάρος μας. Οι συνομιλίε στο Συμβουλίο προχωρούν ικανοποιητικά και πιστεύω ότι εύλογα ο τριμερής διάλογο θα ξεκινήσει με την εκλογή του νέου Κοινοβουλίου. Σήμερα λοιπόν στέλνουμε ένα μήνυμα προς την οικονομία, ότι καταλαβαίνουμε το πρόβλημά τη και ότι είμαστε έτοιμοι να τους προσφέρουμε λύσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Επιτροπέ Μάλμστρεμ. Η κυρία Κράτσα Τσακαροπούλου δεν έχει ακόμα καταφτάσει, γι' αυτό λοιπόν να προτείνω να κάνουμε το εξή, ε, να της δώσουμε πιο πολύ χρόνο ομιλία στο τέλος. Και τώρα να περάσουμε λοιπόν στις, ε, στον κύριο Καλφίν από πλευράς της Επιτροπής ε, Προπολογισμών. Για ένα λεπτό έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή Προπολογισμών θεωρεί ότι η πρόταση για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια είναι εξαιρετική πρόταση, η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια φάση όπου τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε αδυναμία να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Στην Επιτροπή μας διαπιστώσαμε καταρχάς ότι υπάρχει ανάγκη τα κρατημέλη να μην θέσουν επιπλέον όρους στα ΕΜΕΚ, στα συγκεκριμένα δηλαδή κεφάλαια. Επίσης ζητάμε να μην επενδύουν σε παράγωγα προϊόντα. Και τέλος, συμφωνήσαμε ότι πρέπει να λυθούν μέτρα για να μην χρησιμεύουν τα κεφάλαια αυτά στην αποφυγή της φορολογίας. Σας ευχαριστούμε. Συνάδελφε Κάλφιν, τώρα εξ ονόματος των ομάδων, η συνάδελφος κυρία Λουλίν, η οποία είναι εδώ σήμερα μέχρι την τελευταία ημέρα. Και μαζί με την κυρία Κρέστη Γκριλανσμπέγκη έχει μεγάλο ρεκόρ. Μι, μικρόφωνο. Ah. <laughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι για την πρόταση της Επιτροπής και την έκθεση της κυρίας Κράτσα Έχω υποβάλει μια τροπολογία εξ ονόματος της ομάδας μου και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε αμελητή να συνενέσει έτσι ώστε τα επενδυτικά αυτά κεφάλαια να μπορέσουν να ενταχθούν σε άλλα ε, ε, κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τις μακροχρόνιες ε, επενδύσεις και να ενθαρρύνουμε την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Αλλά ας μην αυταπατώμαστε εάν δεν εγγυηθούμε ένα ε, ελάχιστο όρο ευελιξίας δεν θα τα καταφέρουμε. Κάτι το οποίο προτείνω να γίνει μέσω της ε, τροπολογίας μου έτσι ώστε να υπάρχει ένας επιμερισμός με άλλα επενδυτικά εναλλακτικά κεφάλαια ε, επιμένω σε αυτό, διότι έτσι υπάρχει ευελιξία και μείωση κόστους έτσι ώστε τα επενδυτικά αυτά κεφάλαια να ε, προσελκύσουν το ενδιαφέρον για έναν επενδυτή έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει αυτή τη ρευστότητα από ε, το ένα μέρος στο άλλο μέσα στα πλαίσια του, της οικοδόμησης εμπιστοσύνης των επενδυτών και έτσι ώστε και ο μικρός επενδυτής να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία χωρίς υπερβολικά έξοδα. Αυτή η τροπολογία ε, δεν είναι ρήξη και έλευθη, αλλά αποτελεί ένα εχέγγυο και μέσα στα πλαίσια των ΜΕΚ γενικότερα μέσα στα πλαίσια της οδηγίας ε, του 2011 δυνάμει των άρθρων 1, 2 και 49. Όλα αυτά δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα της εποπτείας ε, από τις αρχές ούτε τις ε, προστασίες του επένδυτη. Δείτε το άρθρο 49 της οδηγίας που μιλά για αυτό τα στεγανά στις επενδύσεις, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτές τις ε, επενδύσεις, κάτι το οποίο υποστήριξε και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα αυτή περάσματος των επενδύσεων από τον ένα τομέα στον άλλο χωρίς δυσκολίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα στην συνέχεια τρία λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Ελκαντράουι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπέ, συνάδελφοι, θα ήθελα εξ αρχή ε, ασφαλώ να ευχαριστήσω την καλή συνεργασία για την ε, καλή συνεργασία και για τους συναδέλφους ε, σκιώτε εισηγητές. Θεωρούμε ότι είναι καλή συμφωνία στην οποία καταλήγουμε. σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση τέτοιων μακροπρόθεσμων ε, επενδύσεων. Και αυτέ οι επενδύσει είναι απαραίτητε 100.000 εκατομμύρια έχει. Συγγνώμη, 1.000 εκατομμύρια χρειάζεται η Ευρώπη για να ε, συνεχίσει τις επενδύσεις αυτές και ξέρουμε πόσο γρήγορο δύσκολο είναι σήμερα να γίνουν τραπεζικές ε, χρηματοδοτήσεις και οι αρχές αντιμετωπίζουν προβλήματα και λοιπόν το να κλείσουμε αυτό το χάσμα των επόμενων χρόνων θα είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη πρόκληση και η αξία των επενδύσεων έχει περιοριστεί σε 50% κατά 50% το 2010 και, και τις επόμενα έτη στην Ευρώπη και πρέπει να σας πούμε ότι η επένδυση οι επενδύσεις εξαρτούνται από τραπεζικές πιστώσεις κατά 70% και ξέρουμε ότι οι τράπεζες σφίγγουν τα λουριά για να πληρούν όλες τις ε, κεφαλαιοκές απαιτήσει. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες χρηματοδότησης και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισπανικές, οι ελληνικές και άλλες ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν 33% πιθανότητα να λάβουν ε, χρηματοδότηση. Στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 87% και αυτό τι σημαίνει ότι οι χώρε εκείνε που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα έχουν ακόμα και μεγαλύτερο πρόβλημα επενδύσεων. Τούτου λεχθέντο, αυτό που έχουμε μπροστά μα αποτελεί μια σημαντική προπόθεση για να πληρούνται κάποιοι ποιοτικοί πόροι. Οι νέοι κανόνε σε ό,τι αφορά του δασμικούς επενδυτέ ε, και τη συμμετοχή τους σε διαστατικές επενδύσεις, αλλά δεν ε, μπορούν ε, ανά πάσα στιγμή να αποσύρονται. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι οι επενδυτές θα έχουν συγκεκριμένους ε, πολύ αυστηρούς όρους για να μπορούν να αποσύρουν τα κεφαλαία τους από τις επενδύσεις και θα πρέπει εκ των προτέρων να ανακοινώνονται αυτό, αυτοί οι όροι. Επίσης θα πρέπει να πληρούνται και κάποιοι όροι για το ποια τμήματα σε ποια τμήματα, σε ποια είδη μακροπρόθεσμων τέτοιων ε, προϊόντων μπορεί να γίνονται επενδύσεις ε, σε ό,τι φορά για παράδειγμα τη βιώσιμη ενέργεια, πώς θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των πόρων για να αποφεύγεται ο κίνδυνος, ε, έργα υποδομών τα οποία θα περιγράφονται πιο καλά προκειμένου να μην επενδύουμε σε τομείς που έχουν επαρκή χρηματοδότηση και κλείνοντας είναι σημαντικό να υπάρχουν καμία σύνδεση με φορολογικούς παραδείσους. Εμείς ε, από πλευράς Κοινοβουλίου κάναμε το έργο που μας αναλογούσε. Τώρα το μολάκι πάει στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε Ελμπα Καντράουε. Ο συνάδελφος Πάκρ για 6 λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική πρόταση ενώπιον μας. Μια πρόταση η οποία καθιστά σαφές ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις να έχουν σωστή χρηματοδότηση. Και εγώ πριν από κάνα μήνα έγραψα μια ε, έκθεση, μια ε, έκθεση πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά ακριβώς το θέμα αυτό. Η κρίση λοιπόν Κατά την κρίση η χρηματοδότηση εξαρτώταν βασικά από τις τράπεζες και τώρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τις πηγές χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις αλλά και για τις μακροπρόθεσμα τέτοια διαφορετικά έργα. Απελευθερώνοντας πόρους για να ε, χρηματοδοτούνται αυτά τα έργα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ και επίκαιρη αυτή η πρόταση γιατί θα μπορούσε να δώσει μια όθηση ανάπτυξη και για τις επιχειρήσεις αλλά και για μακροπρόθεσμες, ε, μακροπρόθεσμα επενδυτικά έργα. Περιγράψαμε λοιπόν για ποιου σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ποσοστά και χρήματα αποταμίευσης, κονδύλια αποταμίευσης για μακροπρόθεσμες δεσμεύσει, προκειμένου να φροντίσουμε ότι για παράδειγμα οι επενδύσεις και σε υποδομέ σε δρόμους, σε σιδηροδρόμου, αλλά και σε σχολεία για παράδειγμα θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. Κάναμε λοιπόν κάποιες προβλέψεις που θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση στα κονδύλια αυτά να μην υπάρχει μόνο αυτή η εξάρτηση από τις τράπεζες, αλλά και από τις κεφαλαϊκές αγορές. Αυτό θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση. Θα εξακολουθήσουμε να χρειαζόμαστε και τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει να λάβει πιο πολύ ε, περιθώριο, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να δημιουργηθούν καλύτερες ε, οδοί επενδύσεων. Το νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν προσφέρει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και επενδύσεις για τους fund managers και να υπάρχουν επενδύσεις για διάφορους επενδυτές και μακροπρόθεσμα όραμα. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί μια, ένα νέο κίνητρο στη χρηματοδότηση και διαπιστώνουμε ότι με τις διάφορες νομοθεσίες που ψηφίσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια εδώ στο Κοινοβούλιο που ήταν απαραίτητε για τη σταθερότητα του χρηματοπικονικού συστήματο, είναι πιο δύσκολο για του θεσμικού επενδυτέ να παρέμβουν. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε αυτή την εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε εκ νέου ένα καλό επενδυτικό κλέμα. Πώ οι θεσμικοί επενδυτέ μπορούν να έχουν περιθώριο για να εκπληρώσουν το έργο του, το οποίο είναι η χρηματοδότηση για την επόμενη θετία. Κύριε συνάδελφε Τεπάκερ, σας κάνω σήμα, λέει ο πρόεδρο λίγο, λίγο πιο γρήγορα να μιλάτε, ε, λίγο πιο αργά να μιλάτε, γιατί οι διερμηνεί ε, κάνουν απεγνωσμένες, ε, κάνουν απεγνωσμένα μηνύματα, ότι τρέχετε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Just Μία πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσει το πώς η νομοθεσία αυτή επηρεάζει τους θεσμικούς επενδυτές σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους και τη χρηματοδότησή τους στον αγοράς. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο δίνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η πρόταση να αρχίσει να τονώνει την πραγματική οικονομία και να δημιουργηθούν και θέσεις απασχόλησης, ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ντεμπάκερ. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Φαντάζομαι ότι και οι Ολλανδοί φιλελεύθεροι θέλουν να γίνονται κατανοητοί σε όλη την Ήπειρο και δεν γίνεται αυτό όταν μιλάτε τόσο γρήγορα που δεν σας προφταίνουν οι διερμηνείς. Δεν είναι εδώ ο κύριος Καμάλ, άρα ο λόγος πάει στον κύριο Στόλογιαν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το προσχέδιο ρύθμισης ανταποκρίνεται σε, μια, ε, σε ένα πραγματικό αίτημα της οικονομίας και της αγοράς για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρώπη. Οι τράπεζες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση θέλουν να χρηματοδοτούν μακροπρόθεσμα και να επενδύουν μακροπρόθεσμα διότι έχουν κέρδη βραχυπρόθεσμα. Επίσης υπάρχουν χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα στα οποία δρούν μόνο επαγγελματίες επενδυτές αλλά όπως μπορούν να συμμετάσχουν και οι μικροί επενδυτές, δηλαδή να έχουν αυτή τη δυνατότητα πράγματι και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να πιστεύουν ότι τα ΕΜΕΚ την χάνουν καλής διαχείρισης και προληπτικής διαχείρισης όσον αφορά τη διανομή των κερδών του χαρτοφυλακίου αλλά και του τρόπου τήρησης των κανόνων έτσι ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Η έκθεση περιλαμβάνει τέτοια προληπτικά μέτρα και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Γι' αυτό θα υπερψηφίσω την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Στόλογιαν και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Τόμασίτς για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τα ΕΜΕΚ, είναι οργανισμοί με μακροπρόθεσμους επενδυτικούς στόχους. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν τα κράτη-μέλη. Οι περισσότεροι από εμάς σκέφτονται βραχυπρόθεσμα, δυστυχώς. Πολλά κράτη-μέλη επιπλέον δεν έχουν εθνική στρατηγική στον τομέα αυτών των επενδύσεων. Γι' αυτό και είναι στα πρόθυρα της Οι πολίτες περιμένουν οι ευρωπαϊκές ελίτ να συνειδητοποιήσουν τα σημαντικά αυτά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά Το μόνο που έχουμε στα χέρια μας για μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι τα ΕΜΕΚ. Χρειαζόμαστε όμως για να μπορέσουν να λειτουργήσουν μεταρρυθμίσεις, την δικαιοσύνη, να καταπολεμηθεί η διαφθορά, η χρειαζόμαστε διαφάνεια, άλλη φορολογική πολιτική. Να εγκυμηθουμε λοιπόν ότι έτσι η ευρωπαϊκή οικονομία θα μπορέσει να επανέλθει στο δρόμο της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Τόμα. Έτσι στη διαδικασία ΚΑΣΔΙΑΗ δεν υπάρχει κανένα που έχει ζητήσει το λόγο και γι' αυτό το λόγο θα δώσω στην κυρία Μάλμστρομ. Είμαστε μεταξύ μας πλέον. Λυπική εισηγητρία. Λοιπόν, τα σχόλιά σας θα τα μεταφέρω στον Επίτροπο Μπαρνιέ. Η πρόταση έρχεται με καθυστέρηση, διότι τα ΕΜΕΚ θα δώσουν τη δυνατότητα σε συνταξιδοτικό ταμεία και παρόμοιους επενδυτές να μπορέσουν να επενδύσουν πραγματικά μακροπρόθεσμα. Θα επενδύουν έτσι σε υποδομές, σε έργα τα οποία χρειάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγάλες επενδύσεις και βεβαίω οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις στον τομέα των ακινήτων, ε, μικρομεσαίες και επιχειρήσεις καινοτομίας. Κάτι το οποίο είναι ζωτική σημασία για την εξυγίανση του ψηφιακού τομέα μεταξύ άλλων και για να φέρει ανάπτυξη και θέσει εργασία. Γι' αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο είναι, επαναλαμβάνω, ζωτική σημασία και πρέπει να το θέσουμε στη διάθεση των επιχειρήσεων των συντομότερων δυνατών. Το σημερινό βήμα είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και με την αυριανή σα ψηφορία θα στείλετε και εσεί το μήνυμα ότι η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί προ τη σωστή κατεύθυνση και έτσι σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την αρχή του φθινοπόρου. Ευχαριστώ πολύ και καλό σα βράδυ. Σα ευχαριστώ κυρία Επιτροπή Μάλμστρομ και έτσι λοιπόν ορίστε, ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ε, ψηφοφορία αύριο στις 12. Η... Δημοσιεύτηκε η αυριανή ημερήσια διάταξη για την Ολομέλεια. Σας εύχομαι και σας κύριε Επίτροπε στις ε, υπαλλήλους, στους συναδέλφους και στις